Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Τα, πρακτικά, τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο, οπότε τα πρακτικά εγκρίνονται. Α, για διαδικαστικό ο κύριος Ριμπέρο Κάστρο ε, ζητάει το λόγο. Σας ακούω κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους ε, για λίγα λεπτά που τους κουράζω. Για την